Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να ξεκινήσουμε. Γνωρίζετε ότι θα ξεκινήσουμε με τις αρχαιρεσίες του Προεδρείου για να συγκροτηθούμε σε σώμα. Γι' αυτό και ο Πρόεδρος μας για λίγο έχει εγκαταλείψει θέση του, θα προβούμε πρώτα στην εκλογή του Προέδρου της ομάδας. Διαπιστώνω απαρτία του ενός τετάρτου των μελών, οπότε παρακαλώ ποιος είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου. Ο Σαΐντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα μετά από όριμη σκέψη εννοείται να προτείνω τον κύριο Μπράιαν Σίμψον για τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Άλλοι υποψήφοι υπάρχουν? Όχι. Ο υποψήφιος ε, συμφωνεί. Ε, υποχωρεί. Καλώς διαβοής. Εκλέγεται ο πρόεδρός μας και του παραχωρώ και τον προεδρικό θόκο. Uh, ευχαριστώ που με επανεκλέξατε για τα επόμενα δυόμιση χρόνια ως πρόεδρο. νομίζω ότι δουλέψαμε καλά τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια στην Επιτροπή Μεταφορών και θα συνεχίσουμε και το δεύτερο μισό αυτής της κοινοβουλευτικής εντολής με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι πρόεδρος Επιτροπής αυτής. Και χαίρομαι που ανανεώνετε την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ κύριε Αλκαντράουι που με προτείνατε και σας ευχαριστώ που με εκλέξατε όλους. Πάμε τώρα στο διορισμό των αντιπροέδρων. Διορίζουμε Καταρχήν, τον πρώτο αντιπρόεδρο. Έχουμε τέσσερις αντιπροέδρους. Πάμε λοιπόν στην εκλογή του πρώτου αντιπρόεδρου, του κυρίου Μπός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ρίκια για αντιπρόεδρο. Με προς μεγάλη σας έκπληξη. Ο κύριος Ντομινίκ Ρίκε είναι ο υποψήφιος για πρώτος αντιπρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Μπορούμε να εκλέξουμε διαβοή στον κύριο Ρίκε. Dominic, you'd μπορείς να ανέβεις στο Προεδρείο. Πριν πάμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου, παρακαλώ μπορείτε να στείλετε τους σερβιτόρους εδώ στο Προεδρείο να μας σερβιρούν και εμάς. Τσάι. Πάμε λοιπόν στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου. Ποιοι είναι υποψήφοι για, αυτό το, για αυτή τη θέση. Κυρία Φώστερ. Ο Πίτερ Βαντάλεν είναι η πρότασή μου. Αυτό είναι ο υποψήφιος. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Μπορούμε πάλι διαβοή να εκλέξουμε τον κύριο Βαντάλεν ως δεύτερο αντιπρόεδρο. Συγχαρητήρια, κύριε Βαντάλεν. Πάμε λοιπόν στη θέση του τρίτου αντιπροέδρου τώρα. Κύριε Αλκαντράουι, ποιον έχετε να προτείνετε. Ευχαριστώ. Η Σίλβια Τικάου είναι υποψήφια. Κύριε Τικάου, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για αυτή τη θέση. Μπορούμε να την εκλέξουμε πάλι διαβοής. Sylvia, come and take your place. Μπορείτε να έρθετε και εσείς στο Προεδρείο. Πάμε τώρα στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Κύριε Μπρος. Τον κύριο Κοχ, πρόεδρε, προτείνουμε εμείς. Ο κύριος Κοχ είναι υποψήφιος. Άλλος υποψήφιος υπάρχει? Αν όχι, μπορούμε τον εκλέξουμε διαβοής you'd like to come and join us, we have got room. Δίτερ, σε παρακαλώ, έλα να λάβεις και εσύ θέση στο πεδίο, όσο μένουν άδειες καρέκλες. Okay, now we're going to have to do a little bit of a reshuffle because we've got to get the Polish minister up. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο θέση εδώ γιατί θα έρθει ο Πολωνός Υπουργός. Yeah. Well. Okay, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώσαμε με τις αρχαιρεσίες. Εν συνεχεία πρέπει να υθετήσουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης για τη σημερινή συνεδρίαση. Είστε όλοι ικανοποιημένοι με το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Μπορούμε να εγκρίνουμε επίσης και τα πρακτικά από την, ε, τις 21 με 23 Νοεμβρίου. Τα εγκρίνουμε, όντως. Uh, the 10th well, Και τις 10 Νοεμβρίου. Τα πρακτικά πρέπει να εγκρίνουμε, τα εγκρίναμε όντως και αυτά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας πραγματικό σημείο. Θα ακούσουμε τον ε, Πολωνό Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Νόβακ, ο οποίος θα έρχεται εδώ, για να μας πει τα επιτεύγματα της Πολωνικής Προεδρίας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ και προσωπικά κύριε Πρόεδρε και του συναδέλφου σας για, τη... για τις ε, εκλογές και την συνέχιση τη θητεία σα τα επόμενα δυόμιση χρόνια και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και σας εύχομαι και καλή τύχη και επιτυχία στο υπόλοιπο μισό. Αυτή κανονικά ε, θα είναι η επίσημη ομιλία της πολωνικής κυβέρνησης εκ μέρους πολωνικής προεδρίας και αυτό θα μιλήσω πολωνικά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερο για την ευκαιρία που μου δίνετε ως ε, νέο Υπουργό Μεταφορών ε, ε, ε, Κατασκευών και Οικονομίας της Θάλασσας να σας κάνω μια ανασκόπηση της εξάμηνης Πολωνικής Προεδρίας, του εξαμήνου που πέρασε. Πρώτη την 1η Ιουλίου του προεσμένου έτους η Πολωνία, η Πολωνία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου. Ήταν χαλεπή η πολωνια ανελαβε την προεδρια του συμβουλιου ηταν χαλεπη η καιρη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την, και για την Ευρώπη γενικώ. στο μεταξύ ε, και όσο διεξαγόταν η Προεδρία, η κρίση οξυνόταν όλο και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, η πολωνική κυβέρνηση και η πολωνική κοινωνία με την παραδοσιακή πολωνική αισιοδοξία και την χαρακτηριστική για μας ενέργεια ε, συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας για εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για σύσφυξη της συνεργασίας μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών χωρών. Βέβαια, περισσότερο από πουδήποτε, ο τομέας των μεταφορών είναι αυτό στον οποίο χρειάστηκε ε, να προτάξουμε αυτές τις ε, χαρακτηριστικές ελευθερίες, θεμελιώδεις ελευθερίες, ελεύθερη διακίνηση ε, προσώπων, ε, κυκλοφορία εμπορευμάτων, χαρακτηριστικές ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκεντρώνονται σε αυτό το τομέα που μας ενδιαφέρει όλους, στο τομέα των μεταφορών. Ως νέος υπουργό Μεταφορών θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του προκατόχου μου, του Υπουργού Γκραμπάρτζικ, που σήμερα είναι αντιπρόεδρος ε, της Πολωνικής Βουλής, και θα ήθελα ε, να σας μεταφέρω και τις θερμούς του χαιρετισμού και τις ευχαριστία του για την εξάμεινη συνεργασία, την πολύ αγαστή συνεργασία που είχατε μαζί του. Μου διεμήνυσε να σας μεταφέρω αυτές τις θερμές ευχαριστίες για αυτή την πολύ θετική επαφή που είχατε στο, στη διάρκεια του εξαμήνου η Πολωνική Προεδρία κατάφερε να κάνει πολλά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταφορών. Και νομίζω ότι αφήνουμε ένα πλούσιο κληροδότημα στην διάδοχό μας Δανική Προεδρία, στην οποία και ευχόμαστε φυσικά καλή τύχη. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που μας απασχόλησαν το τελευταίο εξάμεινο. Καταρχήν η Πολωνική Προεδρία ασχολήθηκε με τον κανονισμό για την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Και στις 19 Οκτωβρίου μόλις του προηγούμενου έτους η Προεδρία προέβη σε διεξοδική ανάλυση του κειμένου και ε, εκπώνησε μία συμβαστική πρόταση. Αλλά δυστυχώ είχαμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μα μέχρι τη λήξη Προεδρία και έτσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Γιατί το έγγραφο είναι πολύ σχηδέ και πολύ σύνθετο. Και ε, οι συζητήσει τη 22η Δεκεμβρίου έδειξαν πόσε εκκρεμότητε υπάρχουν και πόση περαιτέρω επεξεργασία χρειάζεται. Γιατί αυτά τα θέματα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών είναι πολύ σημαντικά για τα κράτη-μέλη και οι συζητήσει ήταν αρκετά φορτισμένε συγκινησιακά. Στο ίδιο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, η Πολωνική Προεδρία μαζί με την έκθεση για την πρόοδο των εργασιών υπέβαλε και μία νέα εκδοχή του κειμένου που θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση των εργασιών της Δανικής Προεδρίας. Και θα υποστηρίξουμε φυσικά τους Δανούς φίλους μας ώστε το συντομότερο δυνατόν να διεκπαιρεώσουν το έργο αυτό της αναθεώρησης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία στις εργασίες ό,τι αφορά το πολύ σημαντικό αυτό έγγραφο και ιδιαίτερα να ευχηθώ καλή τύχη στον κύριο Χέρτογκ που είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό γιατί έχει πραγματικά ένα τιτάνιο έργο να επιτελέσει. Πάντως του εύχομαι καλή επιτυχία. Ένα άλλο θέμα που είναι άρκετα συνδεδεμένο με το προηγούμενο αφορά τις διασυνδέσεις των μεταφορών με τις τρίτες χώρες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γείτονες. Και φυσικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε λεωφόρους ε, μεταφορών με τις γειτονικέ χώρες. Και μάλιστα ε, είχαμε τα συμπεράσματα του, Υπουργείου, του Υπουργικού Συμβουλίου Μεταφορών και ένα νέο ε, μια νέα αντίληψη για τις συνεργασίες στις μεταφορές. Είχαμε και ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών των Ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Σχέσης που έγινε το Δεκέμβριο στην Κρακοβία και μάλιστα είχαμε και κοινή δήλωση για τη συνεργασία σε θέματα μεταφορών. Μάλιστα, ένας όρος συνεργασίας σε θέματα μεταφορών με τις γειτονικές χώρες είναι φυσικά η ετοιμότητα των γειτονικών χωρών προκειμένου να εστερνιστούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, κάποια κοινωνικά θέματα, κοινωνικές προδιαγραφές, αλλά και προδιαγραφές ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες ε, σε αυτή τη διάσκεψη, στο άτυπο συμβούλιο με τις χώρες ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης, συμφώνησαν ε, με το θέμα αυτό, όπως αναφέρεται και στην κοινή δήλωση. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την Πολωνική Προεδρία ήταν και το θέμα των θαλάσσιων μεταφορών. Μία από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας ήταν το πρόγραμμα το κοινωνικό πρόγραμμα για τη θάλασσα και μάλιστα το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους είχαμε την πρόταση αναθεώρηση της οδηγίας για το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης των ναυτικών. Και ένα από τα στοιχεία του κοινωνικού προγράμματος για τη θάλασσα ήταν αυτό το θέμα της κατάρτισης των ναυτικών. Το θέμα της κατάρτισης των ναυτικών σχετίζεται άμεσα και με την ασφάλεια στην ναυτιλία και μάλιστα συμφωνήσαμε με τη γενική προσέγγιση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο... φάνηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2011. Γνωρίζω κύριε Πρόεδρε ότι εσείς αναλάβατε και προσωπικά την ευθύνη <laughs> αναλαμβάνοντας την εισήγηση αυτής της έκθεσης και σας εύχομαι καλή τύχη για τη διεκπαιρέωσή της. Η Πολωνική Προεδρία ανέλαβε ε, και την, ε, τις εργασίες για τη δημοσίευση του σχεδίου κανονισμού σε ό,τι αφορά την ε, ταχύτητη κατασκευή για τα δεξαμενόπλια και τα πλοία διπλού τους. Νομίζω ότι αυτό θα μείνει είναι πολύ σημαντικό για το φυσικό περιβάλλον, γιατί πολλές φορές είχαμε ναυάγια με δεξαμενόπλια που οδήγησαν σε πετρελοκυλίδες. Ο στόχος του νέου κανονισμού είναι να αποτρέψουμε και να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί έχουμε πολλές απειλές από πιθανά ναυάγια δεξαμενοπλίων, γι' αυτό και είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί σχετικός κανονισμός για τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους είχαμε τέτοια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο της 22ης Δεκεμβρίου. Η Πολωνική Προεδρία ασχολήθηκε όχι μόνο με τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και με την ολοκληρωμένη πολιτική ε, θαλάσσιων μεταφορών. Και χάρη στις κοινέ προσπάθειες Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταφέραμε να εγκρίνουμε στην πρώτη ανάγνωση τον, τον κανονισμό σε ό,τι φορά την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ε, πολιτική της θάλασσας. Ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο εισηγητής για την έκθεση αυτή, συνέβαλε τα μάλα στην ε, αίσια ε, διεκπαιρέωση αυτού του θέματος, γιατί έδειξε πολύ συνεργάσιμο πνεύμα και τον ευχαριστούμε γιατί ήταν πολύ σημαντική συμβολή του στην ε, υλοποίηση συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την Ευρωπαϊκή Προεδρία ήταν και οι αερομεταφορές. Αφιερώσαμε μεγάλη προσοχή την πρόταση για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες. Το θέμα των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων είναι πολύ σημαντική πρόκληση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την εντολή για την διαπραγμάτευση αεροπορική σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν. Στο ίδιο Συμβούλιο, μάλιστα, ανέλαβε και διαπραγματευτική εντολή ε, για διαπραγματεύσει ψηλού επίπεδου με τη Eurocontrol. Στη διάρκεια τη Πολωνική Προεδρία, ολοκληρώσαμε και τι διαπραγματεύσει ε, τη αεροπορική συμφωνία και με τη Μολδαβία και υπογράψαμε την δήλωση για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρους και την διεύρυνσή του σε τρίτες χώρες στα πλαίσια μιας διάσκεψης που έλαβε χώρα στα τέλη Νοεμβρίου του 2011 στη Βαρσοβία. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την, Ευρωπαϊκή, την Πολωνική Προεδρία ήταν οι χερσαίες μεταφορές. Και στον τομέα αυτό συνεχίσαμε τις προσπάθειες για την αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου και θα ήθελα να αναφέρω ότι ιδιαίτερα για την ε, κυβέρνηση του κυρίου Τούσκ, που έχω την τιμή εδώ να εκπροσωπώ, τα θέματα του εξυγχρονισμού και της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων της Ευρώπης αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Η Πολωνική Προεδρία κατέληξε σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Αυτό συνέβη χάρη στην ε, ε, συμμετοχή και της ε, εισηγητρίας ε, της κυρίας Δέβορα Σαρακιάν και της δικής σα επιτροπής που έδειξε μεγάλη προσήλωση στο θέμα αυτό και χάρη στη δική σας συνεργασία εγκρίθηκαν εγκαίρως οι τροπολογίες, κάτι που επέτρεψε στο Συμβούλιο να καταλήξει στην πολιτική συμφωνία ήδη από το Δεκέμβριο. Φυσικά ευχόμαστε στην Δανική Προεδρία αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό η σχετική οδηγία. Ε, ασχοληθήκαμε και με το θέμα των ταχογράφων, την αναθεώρηση του κανονισμού για τους ταχογράφους και χάρη στην αγαστή συνεργασία ε, καταλήξαμε σε ε, πρώτη συμφωνία για την γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Η Πολωνική Προεδρία όμως δεν ασχολήθηκε μόνο με, μια, με οριζόντια ζητήματα. Είχαμε διάφορες διασκέψεις, σεμινάρια, άτυπες συναντήσεις είχαμε πολλές και διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις ε, που όλες συνέβαλαν ε, πολύ θετικά και νομίζω ότι θα αφήσουν ανεξίτηλα ε, ίχνη και θα επηρεάσουν και τις μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες πτυχές του τομέα των μεταφορών, που είναι και ο τομέας που κατεξοχήν ενδιαφέρει την δική σας Επιτροπή. Και ε, λυπούμε που μακρηγόρησα, έρχομαι εδώ στα συμπεράσματα, στα τελευταία λόγια, αλλά πραγματικά ήταν πολύ εντατικές οι προσπάθειες της Πολωνικής Προεδρίας, γι' αυτό και είχαμε πολλά επιτεύγματα και πολλές συναντήσεις. Πάντως για την Πολωνία που είναι εδώ και 7 χρόνια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή ήταν η πρώτη προεδρία που ασκήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η παρθενική προεδρία ήταν μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την πολωνική κυβέρνηση, αλλά για ολόκληρο τον πολωνικό λαό. Ήταν μια πολύ πλούσια εμπειρία και είμαι πεπισμένος ακράδαντα ότι δεν τα λέω αυτά χάρη ναυρότητας μόνο, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι χάρη στην στενή συνεργασία και την αγαστή συνεργασία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι και εγώ βουλευτή στην Εθνική Βουλή και πραγματικά αναγνωρίζω τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι βουλευτές στη διαμόρφωση της ε, νομοθεσίας και της ε, πολιτικής. Είμαι λοιπόν κράτα πεπισμένο ότι χωρί την αγαστή συνεργασία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα καταφέραμε ω Πολωνική Προεδρία να έχουμε τόσο σημαντικά επιτεύγματα και μάλιστα σε τόσο χαλεπού καιρού και εν μέσω τη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά εκ μέρου τη πολωνική κυβέρνηση και φυσικά εκ μέρου του επιτελείου που με βοήθησε στη και ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά στη διάρκεια τη ε, πολωνική Προεδρίας. Να συγχαρώ θερμά και τον Πρόεδρο και το επόμενο Πρόεδρο, όχι πια ως Προεδρία, αλλά στα πλαίσια του τρίου ε, θα βοηθήσουμε και τη Δανική Προεδρία και την επόμενη Κυπριακή Προεδρία με βάση τις ε, βασικές αρχές που θετήσαμε τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Ελπίζω να κρίνετε και εσείς θετικά την Πολωνική Προεδρία και νομίζω ότι ό,τι καταφέραμε ε, να πετύχουμε θα είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας και για τους διαδόχους μας και πραγματικά πιστεύω στον ε, πολύ ισχυρό ρόλο που θα διαδραματίσει όχι μόνο η Επιτροπή Μεταφορών αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσσωμο για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αποθέτουμε πολύ σοβαρές ελπίδες και προσδοκίες σε αυτή την δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και στη συνέχεια ε, και δεν θα σας πω εις το επανειδήν. Ε, θα βρεθούμε και πριν από την επόμενη Πολωνική Προεδρία που θα γίνει μετά από 14 χρόνια. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πάμε στους συντονιστές τώρα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γκρός Α, συγγνώμη, ο κύριος Ζάντερ πρώτα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό Νόβακ για την εξαιρετική Πολωνική Προεδρία που κατά τη γνώμη των εμπειρογνωμών ήταν από τις καλύτερες ε, ε, προεδρίες των τελευταίων ετών παρόλο που αντιμετώπισε τις αντικσότητες της κρίσης και αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την Πολωνική Προεδρία. Καταφέραμε να υιοθετήσουμε τη γενική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, κατάρτιση των ναυτικών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ε, χαίρομαι που ε, υιοθετήθηκε η μερική προσέγγιση για τα θέματα των ταχογράφων. Νομίζω ότι χάρη στην προσήλωση και την εντατική προσπάθεια της Πολωνικής Προεδρίας, καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο και για το τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ήταν πολύ δύσκολη η πρόοδο, γιατί μόνο στα τέλη του Οκτωβρίου λάβατε το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό δεν κατάφερε η Προεδρία να ασχοληθεί και με το αεροπορικό πακέτο. Ευελπιστώ ότι η Δονική Προεδρία θα δώσει την ιδιαίτερη προσοχή στο πακέτο αυτό. Η περίοδος της ε, Πολωνικής Προεδρίας ήταν πολύ εντατική και για μας, γιατί το τελευταίο εξάμεινο Ολοκληρώσαμε το έγγραφο για την ολοκληρωμένη πολιτική της θάλασσας. Εκφράσαμε τη γνώμη μας ε, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Αερομεταφορών, των Ενιαίων Ευρωπαϊκών Θέρων και είχαμε και την έκθεση ε, Σερατσάνη, τωρικά, στην αναδιατύπωση δηλαδή για το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ ε, και σας ε, και την ΟΚΕ για την ε, συνεδρίαση της 22ης Δεκεμβρίου. Ήταν πολύ σημαντική διάσκεψη αυτή για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς θέρες. Έτσι συνεχίστηκε η Ουγγρική Προεδρία και ελπίζω ότι οι ενιαίοι εθέρες θα αποτελέσουν μία από τις σημαντικές προτεραιότητες και της ευερχόμενης, και της τωρινής μάλλον δανεικής προεδρίας. Στη διάσκεψη της Βαρσοβίας υπόθηκαν όλα όσα έπρεπε να υποθούν. Τέλος ε, τα λόγια λοιπόν πρέπει να περάσουμε στα έργα και να μπορέσουμε εγκαίρως να υιοθετήσουμε τους μεσοπρόθεσμους πόρους ώστε ε, στα τέλη του 2012 να μπούμε σε λειτουργική φάση. Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ την Πολωνική Προεδρία γιατί χάρη σε εσά και χάρη στον προκάτοχό σας, ε, τον κύριο Γκρομπάρτσικ, καταφέραμε να ε, έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία και να υλοποιήσουμε πολλά πράγματα στο τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Αλχαντράουε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της δικής μου ομάδας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Ήταν πραγματικά μια μεταβατική προεδρία γιατί δεν υπήρχαν έτσι μεγάλα θέματα προς ολοκλήρωση. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποιοι φάκελοι οι οποίοι έτυχαν αρκετές, αρκετά καλή διαχείριση και βεβαίως αυτό θα συνεχίσει και τα, επόμενου επόμενους και τα επόμενα χρόνια. Αναφερθήκατε στην κρίση. Όντως και πολύ σωστά το πράξατε. Η πολιτική επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον τομέα των μεταφορών μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και βεβαίως μπορεί να συμβάλλει και στην μελλοντική οικονομική ανάπτυξη για αυτό το πακέτο των διευρωπαϊκών δικτύων. Ξεκινήσατε εσείς τις διαπραγματεύσεις ως προς αυτό και ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες θα υποστηρίξετε την επόμενη Προεδρία, ειδικά όταν μιλούμε για τον προπολογισμό που θα πρέπει να δοθεί για αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, γιατί τα πράγματα θα εξαρτηθούν ακριβώ από τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι. Χρειαζόμαστε τους πόρους για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ε, επενδύσεις και να επιτύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και να δημιουργήσουμε αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και υπάρχει και το Connecting Europe Facility. Η Κομισιόν έχει δώσει ένα αριθμητικό στοιχείο προς αυτό, έχει δώσει τα νούμερα για τον προπολογισμό ελπίζω, για το 2014, ελπίζω ότι θα υπάρξει η στήριξη ως προς αυτό. Και υπάρχει και άλλη μια πτυχή, η οποία νομίζω ότι θα προκύψει στις συζητήσεις που θα κάνουμε με το Συμβούλιο. Και αυτό θα είναι οι συνθήκες. Δηλαδή, κάτω από ποιες συνθήκες ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος μπορεί να τύχει υποστήριξης. Ποιε είναι οι προϋποθέσεις. Εμείς στο παρελθόν είχαμε τονίσει την σημασία τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που έχουν αυτά τα projects και βεβαίως υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν κάποια κριτήρια έτσι ώστε να μπορεί να δίνεται αυτή η στήριξη. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτά τα κριτήρια θα είναι ευρωπαϊκά, ότι θα έχουν μια ευρωπαϊκή πτυχή, μια ευρωπαϊκή διάσταση. Και επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές ναι, κάποια πράγματα έγιναν, προχώρησαν, τα αναφέρατε κι εσείς, ε, μιλήσαμε για την εκπαίδευση των ε, ναυτικών, τα δεξαμενόπλια διπλοκή τους, Μιλήσατε για, την, ε, για τον φάκελο που αφορά την υπηρεσία της θαλάσσιας ασφάλειας, μιλήσατε και για τις αρμοδιότητες που θα έχει. τι θα γίνεται με τη διαχείριση των ε, πλατφορμών για την άντληση πετρελαίου, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα, ατυχήματα κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία. Νομίζω ότι με το φάκελο αυτό κινούμαστε προ σωστή κατεύθυνση και σα ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Να πω επίση ε, για τον Ευρωπαϊκό ε, Εναέριο Χώρο. Έγινε μία διάσκεψη και συζητήθηκε εκεί βεβαίω ο ενιαίος εναέριος ε, χώρο. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχιστεί αυτό να υπάρχει στι ημέρε οι διατάξεις. Βεβαίως πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή από τη θεωρία στην πράξη και αυτό μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εμά μα ανησυχούν λίγο οι προθεσμίες που έχουν τεθεί. Δηλαδή η προθεσμία που υπάρχει για το τέλο του έτου, ε, του τρέχοντο, για τη δημιουργία την, τον, τον μπλοκ αυτό που πρέπει να δημιουργηθούν για τον ενεραίο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να την ε, επιτύχουμε αυτή την προθεσμία εάν δεν λειτουργήσουν όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, εάν δεν αναλάβουν δράση τώρα. Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον ενιαίο ε, ε, εναέριο χώρο, έτσι ώστε να είναι και πιο ασφαλής και βεβαίω αυτό θα ωφελήσει και την ε, βιομηχανία αεροπορικών μεταφορών αλλά και του χρήστε και του πολίτε μα. Νομίζω ότι και εσείς το πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσετε να στηρίζετε όποιε προσπάθειε γίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την εφαρμογή. Όταν θέλουμε να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη πρέπει να έχουμε χρήματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προτεραιότητε έτσι ώστε το 2014 να ξέρουμε τι θα γίνει με τα επιπλέον κονδύλια που χρειαζόμαστε. Όλη η ΡΕΝ επίση έχει ε, παρουσιάσει κάποια πράγματα. Ελπίζουμε αυτά να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα. Επίση, είπατε για τι προτεραιότητε, ε, για τι θαλάσσιε μεταφορέ. Και εμένα βεβαίω ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό και την δική μα την πολιτική ομάδα μα την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίση, η εκπαίδευση των ναυτικών είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε ότι υπάρχει η έλλειψη και ό,τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή του, την κατάρτισή του, τι συνθήκε εργασία του, ε, νομίζω ότι είναι, θα είναι πλεονέκτημα για όλου μα. Γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό στον τομέα αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολλέ νέε θέσει εργασία για νέου και καλοπληρωμένε θέσει εργασία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το προωθήσουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν μια καλή βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Την ΕΜΖΑ επίση θέλουμε να, το, να διευρύνουμε τον φορέα, θέλουμε να αποφεύγουμε ναι, τα ατυχήματα στην, στην θάλασσα. Είδαμε πρόσφατα το ναυάγιο στην Ιταλία. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ε, μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε έτσι ώστε στο μέλλον να αποφεύγουμε τέτοιε μεγάλε κρίσει. Επίση, η θαλάσσια πολιτική. Εγώ είμαι, ήμουν εισηγήτρια πριν προκύψει το νέο, η νέα νομοθετική ε, ρύθμιση και πραγματικά κάνετε πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτό. Κάνατε όντω ε, πολύ καλέ ε, ε, διασκέψει. Ήμουν παρούσα εγώ σε κάποια από αυτές. Χαίρομαι λοιπόν που η θαλάσσια πολιτική ε, πλέον έχει μια νομική βάση και έχει και τίτλο συγκεκριμένο στον ε, προπολογισμό. Αερομεταφορέ. Επίση συμφωνώ, το Single European Sky είναι πολύ σημαντικό, το θέλουμε όλοι. Ε, ξέρω ότι προς το παρόν εξαρτάται από τη Γερμανία και τη Γαλλία περισσότερο και λιγότερο από την Πολωνία, αλλά σίγουρα ότι, ξέρω ότι και εσεί θα συνεχίσετε να προωθείτε τι προσπάθειες αυτέ και στο Συμβούλιο. Είπατε ότι η επόμενη προεδρία σα είναι σε 14 χρόνια. Ε, εντάξει, μπορεί να μην είσαστε εσεί τότε υπουργό, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανεί. Μπορεί να σα ξαναδούμε σε θέση υπουργού. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε πάλι να τα ξαναπούμε και θα βασιστούμε σε όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ εξ ονόματο τη ομάδα μου, τον Υπουργό, Βεβαίω και σε εσά, ε, Πρόεδρε, συγχαρητήρια και ό,τι καλύτερο για την ε, επανεκλογή σα. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω ένα θέμα. Η κοινωνική ατζέντα για του ναυτικού είναι πολύ σημαντική. Για τι θαλάσσιε μεταφορέ βεβαίω υπάρχει και μια οικολογική ατζέντα που είναι επίση πολύ σημαντική. Γιατί οι θαλάσσιε μεταφορέ πραγματικά είναι πολύ ε, σημαντικέ. Μιλούμε για καύση αποβλήτων χωρί φίλτρα αέρο. Μιλούμε για πολύ σημαντικά λοιπόν πράγματα για εκπομπή αερίων ε, που είναι πολύ σημαντική για την για τι θαλασσιέ μεταφορές. Το έχουμε κάνει ήδη σε κάποια ύδατα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και σε πιο ευρύ επίπεδο, ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά για χώρες που έχουν μεγάλες ε, ακτές. Γιατί έτσι αυτό αν δεν γίνει θα καταστραφεί ή θα πληγεί και ο, ο, ε, ο τουρισμός και θα υπάρξει και μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Ε, αυτό που είπε η κυρία Μάισνερ επίση ε, θα συμφωνήσω. Όταν, ε, μόνο όταν έχουμε ατυχήματα και, όταν, και κατόπιν εορτή προσπαθούμε να δράσουμε, πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε από πριν ότι κάτι θα γίνει. Ήδη πριν από 10 χρόνια στο Κοινοβούλιο είχαμε ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, αλλά ελπίζω ότι τώρα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, με τα διπλά κήτη κτλ. τα πράγματα να βελτιωθούν. Επίση, οι αερομεταφορέ. Ε, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον ενιαίο ενέργειο χώρο, αλλά για το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών. Ε, είμαστε αρκετά σκεπτικοί, αλλά εν τω μεταξύ από ό,τι άκουσα, ε, όλες οι αεροπορικές γραμμές που θέλουν να πετούν πάνω από την Ευρώπη δέχτηκαν α, τις προϋποθέσεις αυτού του συστήματος. Θα μπορούσατε να μας πείτε εσείς κάτι γι' αυτό. Ξέρουμε ότι ε, εναντιώνονται στεναρά οι Αμερικανοί, αλλά τώρα αυτό έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε θετική γνώμη. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Επίσης, ε, πολύ θετικό βρίσκω ότι δημιουργείται ένα ε, προηγούμενο, ε, μάλλον αποφεύγεται ένα προηγούμενο με την προσπάθεια της Πολωνίας για αυτά τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν για τις μεταφορές των σιδηροδρόμων. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι α, όταν κάποιο πάρει τόσα πολλά χρήματα ή ένα τομέα πάρει τόσα πολλά χρήματα δεν θα ξέρει τι να τα κάνει. Προφανώ τα ξέρει, αλλά εμεί είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το προέβλεψε αυτό η Πολωνική Προεδρία, γιατί λίγο μετά είχαμε ακριβώ από την ε, Ουγγαρία το ίδιο πρόβλημα. Ήθελαν να μετατρέψουν, να στείλουν τα κονδύλια αυτά σε άλλου ε, κλάδου τα περισσότερα κονδύλια ούτως ή άλλως πηγαίνουν στις ε, χερσαίες μεταφορές. Μόνο 20% πάει στις ε, σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Και χαίρομαι λοιπόν που προέβλεψε η αλλω πηγαινουν στι χερσαιες μεταφορέ, την παει στι σιδηροδρομικες μεταφορέ. και προλάβαμε. Τώρα, για τι ε, κατευθυντήριε γραμμέ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Συζητώνται πολλά και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ξέρουμε ότι η συγκέντρωση σε μεγάλα projects πάει, δεν πάει καλά. Και ξέρουμε ότι οι μεταφορές είναι υπεύθυνε για το 30% των εκπομπών αερίων εμείς θέλουμε να έχουμε και, και μεταφορές μεν, αλλά και καλή προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό δεν γίνεται με μεγάλα project τα οποία θα ολοκληρωθούν σε 30-40 χρόνια και θα καταναλώσουν το 80-90% των ε, κονδυλίων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο γρήγοροι και πρέπει να δούμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είπατε ας πούμε ε, για τη σύνδεση της ε, Βαρσοβίας μέσω του, Πόνς, του Πόσναν από τον Ντάνσικ και μετά προς το Βερολίνο. εντάξει, προς το Βερολίνο προφανώς θα χαρούν πάρα πολύ για τη διασύνδεση αυτή. Χρειάζεται όμω γι' αυτό νομοθετική ρύθμιση. Και το προβλέψατε εσεί στην ε, Πολωνία, ότι το θέμα δεν είναι στα επόμενα ε, δέκα χρόνια να κάνουμε ένα-δυο μεγάλα τέτοια projects, αλλά να γίνει εξυγίανση του υπάρχοντο δικτύου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που το θέσατε ω προτεραιότητα. Το έχουμε και εμεί ω προτεραιότητα και το είχαμε πει και... Ε, και τα προηγούμενα ε, χρόνια προσπαθήσαμε να μειώσουμε την, την, τις χερσαίες μεταφορές και να μεταφέρουμε κάποιο κομμάτι των μεταφορών μας στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. For the ECR, Mr. Van Dalen. Ο κύριος Dalen. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία Κύριε Νόβαξ, ευχαριστώ και εσά και τον προκάτοχό σας, ε, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και με εσά φυσικά. Ήρθε σε επαφή με τι διάφορε πολιτικέ ομάδε για να δει ποιε είναι οι προτεραιότητέ του και για να δει ποια σημεία θα πρέπει να τεθούν στη μερίσια διάταξη προ συζήτηση. Θα ήθελα να μιλήσω για την ε, θαλάσσια πολιτική, γιατί ήμουν εισηγητή και συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με την Προεδρία. Με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό συνεργαστήκαμε και προωθήσαμε πολύ σημαντικά έργα, προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών οργάνων, υπήρχε υπήρχαν διαφορετικές τάσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλαμε να δώσουμε πολλές αρμοδιότητες στην ΕΜΣΑ, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στην Αυσιπλοείας. Εμείς ε, δεν είχαμε διαφωνίες με την Προεδρία και για το Κονκόρτια ε, και για τις ε, ακτές εμείς δείξαμε μεγάλη σύνεση. Πρέπει να δούμε τι συνέβη με αυτό το ατύχημα του υπεροκειάνιου Κονκόρδια. Να μην ξεχνάμε πράγματα όπως η κατάρτιση και να μην ζητάμε κατά ανάγκη κατευθείαν περισσότερη νομοθεσία. Επίσης, για τις, τους πολύτροπους τρόπους μεταφορών. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει το φθινόπωρο του 2011 ότι θα είχε ετοιμάσει ήδη μία νέα πρόταση, αλλά αυτό δεν συνέβη. Θα θέλαμε να είχε δουλέψει περισσότερο η Πολωνική Προεδρία επ' αυτού του θέματος για να, για να το προωθήσουμε. Αλλά τώρα πρέπει απλώς να περιμένουμε. Κύριε Νόβακ, κατά τη συνεργασία με το τρίο των Προεδριών, θα ήθελα να σας ζητήσω να πιέσετε την Κομισιόν για να σπρώξει το θέμα των πολύτροπων μεταφορών. Έχουμε άλλους δύο ομιλητές. Ας τους ακούσουμε. Η κυρία Τικάου πρώτη και μετά θα απαντήσει ο υπουργό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ την Πολωνική Προεδρία ως εισηγήτρια για τον κανονισμό για τους ταχυγράφους, τους ψηφιακούς ταχυγράφους, χαίρομαι για την γενική προσέγγιση που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά τους ψηφιακούς ταχυγράφους. Ξέρω ότι προσπάθησε η Πολωνική Προεδρία να προωθήσει αυτό το θέμα. Ξέρω ότι δεν ασχοληθήκατε με το θέμα της ενσωμάτωσης του χάρτη των ταχυγράφων ή μάλλον του, της κάρτας η οποία θα μπορούσε να προσαρτηθεί στο δίπλωμα οδήγηση. Θα έπρεπε η άδεια οδηγησης και ο κανονισμός για του ταχυγράφους να είναι ένα ενιαίο πακέτο. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ένα δεύτερο θέμα. Γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ που υποστηρίξατε τη θέση των νέων κρατών μελών. Γιατί τα νέα κράτη-μέλη έχουν ε, ανάγκη να αναπτύξουν ε, τις ε, υποδομές μεταφορών τους και ελπίζω αυτές οι ανάγκες να απεικονιστούν σωστά στους διαδρόμους αλλά και στον τρόπο που δίδονται οι χρηματοδοτήσεις για τις ευρωπαϊκές διασυνδέσεις. Ευχαριστώ την ε, Πολωνική Προεδρία. Αυτά που μας είπατε είναι πολύ πλήρη και ευραία. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο κ. Βαντάλεν, ε, που σχολίασε τα θέματα ναυσιπλοείας με πολύ πλήρη τρόπο. Επίσης χαίρομαι για τα σχόλια της Προεδρίας σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών και κυρίως το ΣΕΖΑΡ που θα θα σας επηρεάσει ως Υπουργό. Γιατί εμείς ως Κοινοβούλιο θα πιέσουμε όλες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να κάνουν κάτι πιο επικοδομητικό, ούτως ώστε να προωθήσουμε το ΣΕΖΑΡ. Αυτά που είπε ο κύριος Αλκαντράουι ε, μίλησε για τα Functional Airspace Blocks τα FABs. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη για να προωθηθούν αυτά τα έργα ε, σχετικά με αυτό το θέμα, τα FABs. Θα ήθελα να υποστηρίξετε το θέμα αυτό για να προχωρήσει. Επίσης, τα ωφέλη από το ΣΕΖΑΡ είναι προφανή. Συμφωνήσαμε στην ECR να είμαστε εισηγητές ε, σε μια γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Μα ενδιαφέρει η διαχείριση των ενέργειων μεταφορών, τα θέματα τη τεχνολογία των ενέργειων μεταφορών, όλα αυτά τα πράγματα που θα, υποφε... θα είναι υποφελή για του καταναλωτέ. Θα πιέσουμε λοιπόν στα πλαίσια αυτή τη Επιτροπή και ελπίζω όλοι οι υπουργοί των κρατών μελών να είναι πιο δραστήριοι από ό,τι στο παρελθόν, παρά τι οικονομικέ πιέσει και την οικονομική κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βνόβακ, θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια των Ευρωβουλευτών. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγκάρδια για τα σχόλιά σας και για τις γενικώς πολύ θερμές παρατηρήσεις και πολύ στα σχόλια για την Πολωνική Προεδρία. Ο κύριος ε, Ζασάντε βέβαια ήταν φυσιολογικό είναι να μην είναι αντικειμενικός. Είναι ύποπτος ως προς την υπερβολική ευρώτητα λόγω της ε, καταγωγής του. Είναι Πολωνός, αλλά ε, εκ μέρους του ΕΛΚΑ ευχαριστεί θερμά, την Πολωνική Προεδρία θερμά και τον ευχαριστώ και εγώ και προσωπικά αλλά και εκ μέρους του προκατόχου μου αλλά και εκ μέρους ολόκληρης πολωνική Πολωνικής γιατί πραγματικά εργαστήκαμε πολύ εντατικά και πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα των μεταφορών και για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ελκαντράουι αναφέρθηκε στο Connecting Europe Facility. Αυτός ο μηχανισμός, αυτό το μέσο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας εκ τη πολωνική κυβέρνηση, πια, όχι προεδρία γιατί δεν είμαστε προεδρία, ε, αποδίδουμε ιδιαίτερη σπουδαιότητα και σημασία στο θέμα αυτό και ελπίζω να ε, αφιερωθούν περισσότερα κονδύλια για την ανάπτυξη των υποδομών στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται τέτοιες υποδομές. Και μάλιστα η Πολωνία είναι μία από τις χώρες ε, που αφιερώνει πολλά κονδύλια και κονδύλια συνοχής αλλά και ε, εθνικά κονδύλια προκειμένου να εξυγχρονίσει τις υποδομές ε, στις μεταφορές, χερσές μεταφορές, ε, στις αεροπορικές μεταφορές, σιδηροδρομικές και πιστεύω ότι μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές χάρη και του περιβάλλοντος και να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των υποδομών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο, το Connecting Europe και δεν θα πρέπει φυσικά να δοθεί, να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά και μόνο από το Ταμείο Συνοχής, γιατί θα, θα ήταν αντιφατικό με την ίδια την ιδέα του Ταμείου Συνοχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Μέισνερ, που σημερίζεται τον προβληματισμό μας και για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και για την ΕΜΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Ναυσιπλοείας. Σας ευχαριστώ και για τα θετικά σχόλια που είπατε ε, για τη διοργάνωση των ημερών της θάλασσας που έγινε στη γενέτειρά μου, το Γκδάνσκ. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση και το, αυτή η οργάνωση και για την Πολωνική Προεδρία, αλλά ιδιαίτερα για την πόλη του Γκτάνσκ. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας επισημάνω κάτι που ακούστηκε από πολλούς. Αναφέρθηκε το θλιβερό ναυάγιο που πριν από μία εβδομάδα και κάτι έλαβε χώρα στις ακτές της Ιταλίας, το ναυάγιο του Κώστα Κονκόρντια, του κρουαζιερόπλου. Και φυσικά εκφράσαμε τα συλληπιτήριά μας ε, για αυτή την ε, ε, αποτρόπη τραγωδία που έπληξε την Ιταλία. Και σίγουρα αυτό το ναυάγιο θα συζητηθεί πολύ, συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη, γιατί θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και να καταρτίζουμε όλο και αυστηρότερες προδιαγραφές και να δώσουμε έμφαση και στην κατάρτιση των ναυτικών φυσικά, αλλά και στις προδιαγραφές ε, του εξοπλισμού των κοροαζιεροπλοίων και των ε, πλοίων που πλέον στην Ευρώπη. Ο κύριος Κράμερ μίλησε για την ανάγκη περαιτέρω περιορισμού των καυσέριων και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο των εκπομπών, η πολωνική κυβέρνηση στα πλαίσια της προσπάθειας στήριξης του συστήματος που λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου, εμείς είμαστε θετικοί και θα το υποστηρίξουμε και περαιτέρω. Ο κύριος Κράμερ πριν από λίγο αποκάλυψε το μυστικό μας, γιατί λίγο πριν την σημερινή συνεδρίαση Μιλήσαμε μεταξύ μας για την συνδεση Gdansk Poznań βερολινο Πρόκειται για μια σιδηροδρομική σύνδεση που ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει την έκφαση της ενίσχυσης, της εντατικοποίησης και των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων, γιατί είναι σημαντικές οι αεροπορικές διασυνδέσεις, αλλά δεν, ε, ε, θα πρέπει να μελούμε τις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις και κυρίως ε, τα ταχεία τρένα. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να τα υποστηρίξουμε, τα, τις Ε, Αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα επίση, ε, μια προτεραιότητα της ε, πολωνική Προεδρίας, το θέμα των ε, συνδυασμένων μεταφορών, intermodality. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ το, της διατροπικότητας των συνδυασμένων μεταφορών και θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ε, στην Πολωνία, στη χώρα μου, προκειμένου να προωθηθούν τεχνολογίες που θα ενισχύουν τη διατροπικότητα και θα συμβάλλουν στον καλύτερο συνδυασμό των μεταφορών προκειμένου να αποκομίσουμε και οικονομικό κέρδος αλλά και περιβαλλοντικό όφελος. Ευχαριστώ και την κυρία Τσικάου για τις, για τα, για τις εγκομιαστικές της παρατηρήσεις. Δεν ήταν πρόθεση αυτής της Προεδρίας, γιατί καμία Προεδρία δεν πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τη τα συμφέροντα τη χώρα. Πάει τους πολύ σωστά η κυρία Τσικάου ε, ανέφερε ότι τα θέματα των διαδρόμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών αλλά και για τα ενισχυμένα αυτά τα γενικότερα δίκτυα το θέμα των υποδομών και των διαδρόμων είναι πολύ σημαντικά και για την Πολωνία. Και καλό θα ήταν να φτάσουμε σε αυτό το τρίτο επίπεδο και σίγουρα δεν θα πρέπει η συνέχιση να γίνει εις βάρος ε, των ε, ήδη συμπεφωνηθέντων για τα 10T. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Φώστερ, είμαστε υπέρ των FABs και σίγουρα ε, ετοιμαζόμαστε και η Πολωνία ασχολείται με τα FABs και ετοιμάζει FABs με τη γειτονική Λιθουανία. Θέλουμε φυσικά να ενισχύσουμε τα συστήματα που θα βελτιώσουν και την ποιότητα και την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και την, θα βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών προς τους συμπολίτε μας στα πλαίσια και των κοινών ευρωπαϊκών εθέρων. Όλα αυτά τα θέματα που ήταν προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητες της πολωνικής κυβέρνησης. Και όλα αυτά που πράξαμε το προηγούμενο εξάμενο δεν ήταν αντιφατικά με τις προτεραιότητες και της ε, πολωνικής κυβέρνησης, γιατί η Πολωνία θεωρεί ότι είναι απόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που θα εμβαθύνουν την, ε, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι προς το συμφέρον όλων μας και της Πολωνίας. Αυτά. Αυτά ως προς τις ε, συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ευελπιστώ ότι θα είναι αυτή η τελευταία μας συνάντηση. Προσβλέπω σε συνέχιση της ε, στενής συνεργασίας και της αγαστής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ακράδαντα στον ιδιαίτερο ρόλο που θα διδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης αυτής. Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί εδώ χτυπά ο παλμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη προ το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευχαριστώ θερμά και καλή τύχη στου διαδόχου μα στη Δανική Προεδρία. Μπορεί να υπολογίζει και στη δική μα υποστήριξη φυσικά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλή τύχη και στο Υπουργείο σας. Τώρα θα συνεργαστείτε στα πλαίσια της Τρόικας με τους Δανούς και τους Κύπριους. Και θα σήμουν ευγνώμων αν εκφράσετε και τις ευχαριστίες σας, τις ευχαριστίες μας μάλλον, στον προκάτοχό σας που είναι τώρα α, αντιπρόεδρος της Βουλής. Τον ευχαριστούμε και αυτόν. Ε, προσβλέπουμε στην ε, συνεργασία μαζί σας σε αυτές τις άτυπες συναντήσεις του Συμβουλίου που λαμβάνουν χώρα από καιρούς καιρών. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να μας κάνετε αυτή την παρουσίαση. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών μέχρι τις 4 και 4, περιμένοντας την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Σομπιεράσκα. Δώστε μου 10 λεπτά για να αρχίσω να ψελίζω σωστά, να μάθω να ψελίζω σωστά το όνομα της α, Υπουργού. 10 λεπτά διάλειμμα λοιπόν. Ωραία. Okay, on the Ωραία, συνάδελφοι. Λίγοι μείναμε, αλλά αυτοί που έχουν σημασία είναι εδώ. Οπότε να περάσουμε στο επόμενο σημείο για την ανταλλαγή απόψεων με την Πολωνή Υπουργό. Ελπίζω το όνομά σας να μην το σκότωσα εντελώς. Αν το σκότωσα, σας ζητώ συγγνώμη. Θα δούμε τα θέματα τουρισμού Βεβαίω και κατά τη διάρκεια των όσων έγιναν στην ε, Πολωνική Προεδρία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έρχομαι και πάλι στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας παρουσιάσω σημαντικά επιτεύγματα της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου στα θέματα του τουρισμού φυσικά. Θα ήθελα να πω ότι η Πολωνική Προεδρία ε, διεξήχθη σε μια δύσκολη στιγμή, σε χαλεπούς καιρούς, σε καιρούς που αποτελούσαν ακόμη, απαιτούσαν ακόμη μεγαλύτερη και βαθύτερη συνεργασία και ε, άρα ε, αντιμετώπιση πολύ σημαντικότερων προκλήσεων. Και μάλιστα η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη περισσότερο ήταν στραμμένη στο θέμα της διασφάλισης της ε, χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας της Ευρωζώνης. Και επικεντρώθηκε σε οικονομικούς τομείς που μπορούσαν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και ένας τέτοιος τομέας ακριβώς είναι ο τουρισμός που μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ήδη από την έναρξη της Προεδρίας τον Ιούλιο σας ανέφερα ότι ο τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το θέμα της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού ε, γι' αυτό σκοπεύαμε να κάνουμε μια διάγνωση και να προβούμε σε κάποιες συστάσεις. Αυτή ήταν ε, η πρώτη φυσικά προεδρία της Πολωνίας στο Συμβούλιο και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική και εμπειρία, αλλά πολύ σημαντική και πρόκληση. Οι προτεραιότητες που προτείναμε ε, απέρευσαν και από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, προέβλεπε το νέο πλαίσιο της πολιτικής τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχε άμεση σχέση και με τις προτεραιότητες της στρατηγικής ε, του 2020. Μάλιστα στο θέμα αυτό ε, αφιερώσαμε και τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Πολωνικής Προεδρίας για τα θέματα τουρισμού. Δηλαδή συνδιοργανώσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού που έλαβε χώρα στις 5 έως 7 Οκτωβρίου στην Κρακοβία και το κυρίως θέμα αυτού του φόρουμ ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον ευρωπαϊκό τομέα του τουρισμού. Πέραν της ολομέλειας ε, του φόρουμ είχαμε και δύο ξεχωριστά πάνελ εμπειρογνωμόνων. Το πρώτο πάνελ ασχολήθηκε με την εμπέδωση των βάσεων και της επιστημονικής και κοινωνικής γνώσης ό,τι αφορά τον τουρισμό και το δεύτερο πάνελ αφιερώθηκε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα στην καινοτομία και στην τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας στο θέμα του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά το πρώτο πάνελ των εμπειρογνωμόνων, που όπως σας είπα αφιερώθηκε στη, στις βάσεις ε, της επιστημονικής και κοινωνικής γνώμης. τα συμπεράσματα που απέρευσαν από τη συζήτηση στο πάνελ αυτό έτειναν προς την ανάγκη ε, διάδοσης της γνώσης σε διάφορους ε, τομείς, σε διάφορες ομάδες επιστημονικές και κοινωνικές για να δημιουργηθεί καλύτερη γνώση για το θέμα του τουρισμού. Και μάλιστα ε, θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία μιας βάσης που θα συγκεντρώνει την ευρεία γνώση που αφορά όλες τις τάσεις ε, που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Και δεν ε, ε, περιλαμβάνονται εδώ μόνο στατιστικά δεδομένα, αλλά και δεδομένα marketing, αναλύσεις για τις δημογραφικές τάσεις και επίσης και πληροφορίες ε, για συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές του τουρισμού. Αυτά τα δεδομένα και κυρίως τα δεδομένα που, που αφορούν τις αναλύσεις και την αξιολόγηση συγκεκριμένων οικονομικών ε, ε, τάσεων έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους ενδιαφερομένους του κλάδου, αλλά κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σε ένα ενιαίο μέρος, σε μια ενιαία βάση, διευκολύνεται καλύτερα το έργο τους και μπορούν καλύτερα να προγραμματίσουν ε, τα επιχειρηματικά του σχέδια και τη δραστηριότητές της. Γι' αυτό και προτείναμε τη δημιουργία ενός εικονικού ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου του τουρισμού, κάτι που περιλαμβάνεται και στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η η Ιταλική εμπειρία, το Ιταλικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε στο φόρουμ, ε, έδειξε ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, δημιουργώντας διάφορες στρατηγικές ανάπτυξης του τουρισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Φέτος, περιμένουμε στον τομέα του τουρισμού συγκεκριμένες δραστηριότητες γιατί το σχέδιο εργασιών για το 2012 στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της κοινοτομίας προβλέπει την χρηματοδότηση της έναρξης των εργασιών για τον τομέα αυτό και μάλιστα χρηματοδότηση κυρίως ε, του έργου των ε, εμπειρογνωμόνων προκειμένου να εντοπιστούν κάποια κενά ε, σε ό,τι αφορά τις έρευνες ε, του μάρκετινγκ ε, και τις οικονομικές έρευνες που είναι προσιτές. Επίσης, σημαντικό θέμα είναι η συνεργασία με τον ΟΣΑ και άλλες διεθνείς οργανώσεις, η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού, για παράδειγμα. Εδώ και πολλά χρόνια οι οργανισμοί αυτοί έχουν πολύ άριθμες δραστηριότητες και με δορυφορικά εργαλεία μπορούν να αναλύσουν διάφορες ε, τάσεις και ευρωπαϊκές και παγκόσμιες. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των προσπαθειών θα λάβει χώρα και η οριστικοποίηση, η ολοκλήρωση μάλλον των ε, κρεμών ερευνών και στόχο ε, έχουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο πόρταλ του ίντερνετ και μια ενιαία βάση που θα είναι προσιτή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεύτερο ζήτημα που εξετάστηκε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ του Τουρισμού ήταν, όπως σας είπα, η καινοτομία και οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας για τον τουρισμό πάντα. Η, η οικονομική ύφεση φυσικά επηρεάζει αρνητικά την, τον τουρισμό όπως και τους άλλους οικονομικούς κλάδους. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στον τουρισμό. Μας ενδιαφέρουν φυσικά οι καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στον τουρισμό, αλλά δεν αποτελούν πάντα εχέγγυα για τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών προϊόντων. Από τη συζήτηση που έγινε στο φόρουμ, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γενικευθεί φυσικά η δυνατότητα χρήσης τέτοιων ε, τεχνολογιών σε ε, όλο το φάσμα του τουριστικού κλάδου. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που δείχνουν ότι η χρήση τέτοιων τεχνολογιών εξυγχρονίζει την ευρωπαϊκή προσφορά στον τουρισμό, αλλά με πολύ σημαντικό ε, τρόπο ταυτόχρονα εξορθολογίζει και το κόστος της δαπάνες ε, αυτής της προσφοράς στον τουρισμό. Αναφέρθηκα προηγουμένως και στο, στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που προβλέπεται για το 2012 και δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα από τη συζήτηση στο φόρουμ προέκυψε ότι τα τουριστικά σχέδια που χρησιμοποιούν την καινοτομία, που αξιοποιούν την καινοτομία, ε, αξίζουν και κάποιες οικονομικής υποστήριξης και είναι επιλέξιμα και οικονομική υποστήριξη και χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιολογώντας τώρα τα αποτελέσματα αυτού του Ευρωπαϊκού Φόρουμ του Τουρισμού στην ε, Κρακοβία, θα πρέπει να αναφερθούμε και στις εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο και ε, στο περιθώριο αυτού του φόρουμ Έγιναν, για παράδειγμα, κάποιες συναντήσεις ε, των περιφερειών της Ευρώπης και έγινε μια, η παρουσίαση μιας πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλίας του διοντολογικού κώδικα ή του κώδικα ε, βέλτιστων πρακτικών ε, για τον αηφόρο τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες. Η αηφόρος ανάπτυξη του τουρισμού είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της νέας ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Τουρισμού. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε και να διαδώσουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ο κώδικας αυτό των καλών πρακτικών καταρτίστηκε κυρίως ε, για, τη χρήση, για χρήση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα τον ε, αισθενιστούν οικειοθελώς. Το, στο σχέδιο ε, εκπόνηση αυτού του ε, κώδικα συμμετείχαν δύο επιστημονικοί κλάδοι και πέντε ε, πολωνικές εταιρείες καθώς και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Αυτό το σχέδιο του κώδικα βρίσκεται στην τελική του φάση, δηλαδή στην φάση της προαιρετικής ε, υιοθέτησή του από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ε, και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμότατα τον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπή Μεταφορά και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κάρλο Φιντάντσα, για, πολύ, για την πολύ ενεργό συμμετοχή του στο Φόρουμ του Τουρισμού. που μας παρουσίασε την ε, προσέγγιση της ε, δικής της Επιτροπής ό,τι αφορά τις διάφορες προτάσεις για τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ένα, μια άλλη εκδήλωση που έγινε ε, στα παράλληλα με το φόρουμ ήταν το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού. το, άτυπο αυτό Συμβούλιο έγινε το Δεκέμβριο, όπως και το φόρουμ αυτό στην Κρακοβία και θέμα του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού ήταν η προαγωγή της Ευρώπης ε, ως σημαντικού τουριστικού προορισμού και η πρόθεση αυτή κυρίως σε εξωευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες BRIC. Οι συζητήσει σε αυτό το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού έδειξαν ότι τα κράτη-μέλη γενικώ είναι υπέρ αυτής της κατεύθυνση ε, των εργασιών που κατά τη γνώμη μα ε, έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα μια στιγμή που διαπιστώνουμε μια οικονομική επιβράδυνση γιατί στα πλαίσια της οικονομικής επιβράδυσης αποδυναμώθηκε και ο τουρισμός. Οποιαδήποτε λοιπόν δράση και εργασία μπορεί να βελτιώσει τον τουρισμό και να ενισχύσει τον τουρισμό προς την Ευρώπη έχει σημασία. Με την έγκριση αυτών των πρωτοβουλειών ε, και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Υπουργοί μίλησαν και για την ε, ανάγκη φυσικά τήρησης της αρχής επικουρικότητας. Όπως είπα όμως, αυτή η εντατικοποίηση των εργασιών προκειμένου να προαχθεί η Ευρώπη σε τρίτες αγορές ως τουριστικός προορισμός χρήζει ευρυθέστερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ε, κρατών μελών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού και των εθνικών ε, αντίστοιχων τουρισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού έχει φυσικά πλούσια εμπειρία σε θέματα προαγωγής της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού στις τρίτες χώρες. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι στα πλαίσια του άτυπου συμβουλίου στην Κρακοβία καταφέραμε και υπογράψαμε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού με βάση την οποία θα προωθηθούν ε, ταξίδια προς την Ευρώπη με το σύνθημα ε, «Η Ευρώπη το ατέρμονο ταξίδι». Ε, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν το υπάρχον πορτάλ, το visiteurope.com και ξεκίνησαν και κάποιες διαφημίσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι ξέρω, ήδη την 1η Δεκεμβρίου του 2011 έγιναν τέτοιες διαφημιστικές εκστρατείες υπέρ της Ευρώπης τουριστικού τουρισμού στην Κινέζικη αγορά. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών έγινε λόγος φυσικά για αυτή την προαγωγή της Ευρώπης στις τρίτες αγορές αλλά δεν αναφέρθηκε το θέμα των θεωρήσεων. Θυμάμαι την συζήτηση που είχαμε τον Ιούλιο και ε, σε εκείνη τη συζήτηση αναφέρθηκε το θέμα των θεωρήσεων, γιατί η Πολωνία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στα πλαίσια φυσικά των ε, νομικών δυνατοτήτων μας να ε, απλουστευτούν στο μέγιστο οι οι διαδικασίε ε, χορήγηση θεώρηση, ιδιαίτερα για υπηκόου τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να υλοποιήσουμε τη μεγαλεπίβολη πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή, που είναι το σχέδιο για 50.000 τουρίστες, δηλαδή για τις τουριστικές ανταλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιού Αμερικής. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη Χιλή ε, σε περιόδους που είναι εκτός των περιόδων τουριστικής εχμής και γι' αυτό το θέμα των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε συμφέρον στο μέτρο των δυνατοτήτων ε, οι διατυπώσεις για τη χωρίς θεωρήσεων είναι όσο πιο απλές γίνονται. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που παρουσιάστηκε στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο και που μίλησε για την σύσταση ειδική ομάδα εργασία που θα ασχοληθεί με την απλούστευση αυτών των διατυπώσεων για τι θεωρήσει. Επαναλαμβάνω, έχουμε πρόταση για τουριστικές ανταλλαγές με τη Βραζιλία και η Βραζιλία δήλωσε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την τουριστική προσφορά της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε την πολύ ισχυρή προσφορά, τουριστική προσφορά των Αμερικανών, ε, των Βόρειο Αμερικανών στην ε, αγορά της Λατινικής Αμερικής. Επαναλαμβάνω, ο αηφόρος τουρισμός είναι σημαντική προτεραιότητα της Πολωνίας και αποτελεί και την προτεραιότητα της ανακοίνωσης. Η Πολωνία θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων αυτής της ανακοίνωσης και μάλιστα το Δεκέμβριο, σχετικά πρόσφατα, 7 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, από κοινού με, τις, ε, με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ε, για τους, ε, των ποδηλατών. Ε, ασχοληθήκαμε με τις, τα ευρωπαϊκά ποδηλατικά μονοπάτια και Είχαμε και το νέο μονοπάτι 13, το μονοπάτι του σιδηρού παραπεδάσματος και μιλήσαμε και για την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία περαιτέρω ποδηλατικών μονοπατιών. Τώρα, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση να εκφράσω την ικανοποίησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το προηγούμενο Δεκέμβριο του ψηφίσματος για, το Ευρωπαϊκό, για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών μετά από πρόταση της δικής σας Επιτροπής και εκεί υπάρχει η έκκληση για να συμπεριληφθούν και οι τα μονοπάτια, τα ποδηλατικά, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Αυτή η έκκληση για μας έχει μεγάλη σημασία και συμβάλλει στην αηφόρο, ε, στην αηφόρο ανάπτυξη όχι μόνο των μεταφορών, αλλά και του τουρισμού. Και τελικά, σε τελική ανάλυση, ερχόμαστε στο θέμα της χρηματοδότησης, που είναι και το πιο σημαντικό, γιατί έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές για το 2013-2020, την επόμενη επταετία, έχοντας επίγνωση της δυσκολίες της κατάστασης. Στα πλαίσια του τρίου η Πολωνία θα ε, βοηθήσει και τη Δανική και την Κυπριακή Προεδρία προκειμένου να αναζητήσουν τις κατάλληλες ε, συμβιβαστικές λύσεις ε, για να στηρίξουμε τον τουρισμό, γιατί ιδιαίτερα σε αυτή την χαλεπή περίοδο για την οικονομία, χάρη στον τουρισμό μπορούμε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Κατά την κατάρτιση αυτών των νέων δημοσιονομικών προπτικών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στα πλαίσια των ισχυών των περιορισμών να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί ο τουρισμός είναι ένας οριζόντιος κλάδος και η ανάπτυξή του ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και άλλων τομέων. Οπότε η χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, στον τουρισμό θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της προσφοράς και σε άλλους τομείς. Και, στην, και στον τομέα αυτό προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία και στην υποστήριξη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού συνάδουν με τα συμπεράσματα της Πολωνικής Προεδρίας που παρουσιάστηκαν ε, το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή που μου δώσατε. Είμαι στη διάθεσή σας σε περίπτωση που υπάρχουν ε, απορίες, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, for that very... Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την πλήρη σας αυτή παρουσίαση. Για πρώτη φορά βλέπω τον κύριο Κράμερ να χαμογελάει. Και όταν αναφέρατε αυτά τα μονοπάτια του συντρού παραπετάσματος, που όλοι γνωρίζουμε, θα ε, καταφατικά. Ο κύριος Γκρός από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό, εξ ονόματος ε, του ΕΛΚ. Χαίρομαι που είχατε αναλάβει την Προεδρία την, και την ολοκληρώσατε με μεγάλη επιτυχία. Έπρεπε καταρχά να συντονιστούμε πριν μπορέσουμε να νομοθετήσουμε. Νομίζω ότι για, αυτό, για αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της εργασίας σας. Και Τώρα, αυτή αν ήταν άτυπη αυτή η συνάντηση των Υπουργών ή αν ήταν το φόρουμ ε, που βοήθησε, νομίζω ότι και τα δύο ήταν πολύ θετικά και έδειξαν την συνεργασία που είχατε δηλώσει ότι θέλετε να έχετε με το ε, Κοινοβούλιο. Και τελικά το πετύχατε. Για τον τουρισμό. Είπατε κι εσείς ότι και για εμάς είναι ένας τομέας αυτός που θα καλύψει, θα φάει μάλλον πολύ χρόνο από το Κοινοβούλιο, γιατί ο τουρισμός έχει τόσες πολλές πτυχές, είναι πολύ σχηδής τομέας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο συντονισμός λοιπόν και εδώ εσωτερικά στο Κοινοβούλιο είναι σημαντικός, ε, είτε μιλάμε για κοινωνική πολιτική, είτε για περιφερειακή πολιτική, είτε για πολιτική κινητικότητας για την κινητικότητα ε, υπεύθυνε είναι οι μεταφορέ. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα μα απασχολήσει για πολύ καιρό. Ο τουρισμό, ε, ίσω σε κάποιε περιφέρειε, να είναι και ο δεύτερο ή ο τρίτο πόρο ε, εσόδων. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μα. Ελπίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι στα πλαίσια τη κινητικότητα θα υπάρξει μια έτσι συλλεκτική, μια γέφυρα, σύνδεση μεταξύ των ε, στόχων που έχουμε θέσει για τις μεταφορές του αύριο αλλά και για τον τουρισμό. Ε, δηλαδή η χρήση των ε, θαλασσιών οδών, για των μονοπατιών των ποδηλατών, δεν θα τα πω, φαντάζομαι ότι θα τα πει ο κύριος Κράμερ αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι στόχοι, κάποια σημεία στα οποία νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε κυρίως τον τουρισμό και την κινητικότητα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ε, μεγάλο εύρος και πεδίο δράσης εδώ. Ε, ο πρόεδρος το είχε πει και πιο πριν ότι και η ιστορία και ο πολιτισμός και η φύση είναι κληρονομιά ε, που θα πρέπει ο τουρισμός όχι μόνο να την καλύψει αλλά και να την προωθήσει, να την παρουσιάσει, να την αναδείξει. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν και οι απαραίτητοι πόροι για να γίνουν όλα αυτά. Στον τομέα αυτό επίσης δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν και αύριο οι επιχειρήσει αυτέ, να χρησιμοποιήσουμε τι ε, γραμμέ του προπολογισμού, όχι για να δημιουργήσουμε νέε δομέ, αλλά για να βοηθήσουμε αυτέ τι μικρέ και μεσαίε δομέ που υπάρχουν, να δώσουμε σε αυτέ τι επιχειρήσει πρόσβαση, σε πληροφορίες, ε, σε δίκτυα, σε πόρου, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό περιμένουμε. Εμεί, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δέσμευση που δείξατε κατά τη διάρκεια της προεδρία σα και ελπίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο, προ... ο θα λάβει τη θέση που του εφαρμόζει και στο Κοινοβούλιο, όπω έκανε και στα πλαίσια τη Προεδρία σα, σε όλε τι πτυχέ τη πολιτική και τη κοινωνική πολιτική και τη οικονομική. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ε, εικόνα που θα δίδεται προ τα έξω, ε, σεβόμενη πάντα και την ε, πολυπλοκότητα των διαφόρων περιφερειών. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα. Ο ο κ. Αλκαντράουι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την πολύ πλήρη εισαγωγή σας. Δεν μείνατε με σταυρωμένα χέρια, αυτό φαίνεται. Αντίθετα, εμείς δεν μπορώ να πω ότι δουλέψαμε εργοδός υπέρ του τουρισμού. Από την εισαγωγή σας προκύπτει όμως ότι ο τουρισμός έχει πολλές πτυχές, πολλές πλευρές και για τις μεταφορές, για τα δικαιώματα των επιβατών, για τις υποδομές, Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ε, τομέων αυτών και του τουρισμού. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μια σφαιρική, μια ενιαία προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τον εναρμονισμό των, χρησ... των κριτηρίων ποιότητας του label, εμείς πουλάμε την μάρκα Ευρώπη. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ποικιλομορφία σε τουριστικό επίπεδο στην Ευρώπη και θα μπορούσαμε, ε, αν συνεργαζόμαστε, να κάνουμε τεράστιες οικονομίες κλίμακας. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναλυθεί πολλές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό στον τουρισμό που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί και νομίζω ε, θα πρέπει να επιταχύνουμε λιγάκι τις προσπάθειές μας. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο έχει ετοιμάσει μια πολύ σημαντική έκθεση πρωτοβουλίας με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που δεν θα σα απαριθμίσω εδώ, αλλά μέσα στο 2012 θα γίνει κάτι σημαντικό. Θα πρέπει να πείσουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν να προβλέψουν ένα, μια γραμμή στον προϋπολογισμό για τον τουρισμό στα πλαίσια των, των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020. Θα ήταν ένα πρώτο βήμα, ούτως ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική τουρισμού. Ξέρω ότι οι περιφέρειες, οι χώρες, οι πόλες εξαρτώνται ακόμα από τις δικές τους πολιτικές, αλλά θα πρέπει να πείσουμε αυτές τις περιοχές, αυτές τις πόλεις, ότι αν συνεργαστούμε, αν δουλέψουμε μαζί, θα έχουμε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα και θα κερδίσουν όλοι. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, τη χωριστή γραμμή προπολογισμού για τον τουρισμό. Εμεί ε, το θέλουμε στο Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε μια σειρά από πρωτοβουλίε. Μιλήσαμε για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά υπάρχουν και άλλε πρωτοβουλίε που προωθεί το Κοινοβούλιο. Για να καταλήξω, Σα ευχαριστώ ακόμα κυρία Υπουργέ για τη δουλειά σα, για την προσπάθειά σα και μαζί με εσά και τους διαδόχους σας θα δώσουμε στον τουρισμό τη θέση που του αρμόζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τους φιλελεύθερους. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ε, συγχαίρω για την εκλογή σας. Ε, θέλω να συγχαρώ και την κυρία Υπουργό για την δεσμευσή της, για το πάθος, για τη ζέση που έδειξε αυτό το εξάμεινο για να προωθήσει διάφορα θέματα που για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νέα. Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας πέρυσι, εμείς είχαμε μια πολύ έντονη περίοδο στην προσπάθεια να συγκεκριμενοποιήσουμε και να δώσουμε σάρκα και οστά σε ένα άρθρο που έδινε απλώ κάποιε δυνατότητε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια στη Μαδρίτη με την Ισπανική Προεδρία, με τη συνάντηση των ενδιαφερομένων, των stakeholders. Συνεχίσαμε με τη δική σας ε, Προεδρία ε, και όπως ακριβώ είπαν και οι συνάδελφοι, ε, ο φάκελος που πρόθεσε η Επιτροπή μα ήταν, το θέμα μάλλον που πρόθεσε η Επιτροπή μα ήταν η χρηματοδότηση και αυτή ήταν η βάση για να δουλέψουμε. Υπάρχει πολύ δυναμικό εδώ που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για να μην υπάρξει ο κίνδυνος, όταν έχουμε τόσα εργαλεία στη διάθεσή μας, τόσα ε, μέσα, τα ξεχνάμε και ψάχνουμε να βρούμε νέα ή να φτιάξουμε νέα ε, και ένα νέο προγραμματισμό. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κίνδυνος, θέλουμε να τον αποφύγουμε. Γι' αυτό σας θέτω το εξή ερώτημα. Τι όρια υπάρχουν σε αυτό το φάκελο που εκπώνησε το Κοινοβούλιο και τι όρια βρήκε η Πολωνική Προεδρία για να περιορίσει και το χρόνο. Έξι μήνες δεν αρκούν για να προωθήσουμε θέματα τόσο σημαντικά. Δηλαδή, τι, ήταν αυτό, ποια ήταν τα εμπόδια, να το πω καλύτερα, που δημιούργησαν πρόβλημα στην ε, Πολωνική Προεδρία. Ακούσαμε από την Υπουργό σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν εντοπιστεί κάποιες προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Έγινε αυτό το workshop στο Dansk και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε και ο κύριος Αλκαντράουι, νομίζω ότι σύντομα θα πρέπει στην Επιτροπή να πάει αυτό το κείμενο, ούτω ώστε να εξετάσουμε πώς ε, ο οικονομικός προγραμματισμός, η χρηματοδότηση δηλαδή, θα προωθηθεί και ποιες διορθωτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να επιφέρουμε, ούτω ώστε να αρχίσουμε πραγματικά να απτύσσουμε το δυναμικό του τουρισμού μέσα στην οικονομική συγκυρία μας. Ευχαριστώ, κύριο Κράμερ. Και εγώ να ευχαριστήσω την Υπουργό για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, αλλά και πιο πριν. Θα θυμάμαι πολλές ε, συναντήσεις που είχαμε στην Μαδρίτη για την προετοιμασία. Ελπίζω ότι και στο μέλλον η συνεργασία μας θα παραμείνει αγαστή. Και από την δική μου πλευρά, Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Υπουργό Οι υπουργοί λένε στη Γερμανία μπορούν να αλλάζουν ε, αρκεί οι γενικοί γραμματείς να παραμένουν στις θέσεις τους ε, και νομίζω ότι παρόλο που άλλαξε καθήκοντα υπουργό, ε, θα συνεχίσει να εργάζεται πολύ καλά. Μιλήσατε για τον, για τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός τομέας. Υπάρχουν πολλά αρνητικά παραδείγματα που μπορούν να τον πλήξουν. Δεν χρειάζεται όμως να επαναλαμβάνουμε τα αρνητικά, μόνο τα θετικά. θα... Και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με την αναθεώρηση θεώρηση του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υποθέτω ότι και εσεί θα δεσμευτείτε έτσι ώστε και αυτά τα ταμεία να συνδεθούν με τον α, τουρισμό. Υπάρχουν κάποια αριθμητικά στοιχεία, κάποιε γραμμές του προπολογισμού για τα μεγάλα projects, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά για τα μικρά δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να μιλούμε για α, βιώσιμο τουρισμό θα πρέπει να υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ε, δημοσιονομικό, στον προπολογισμό, γιατί πραγματικά έτσι θα δοθεί μεγαλύτερη όθηση. Και αυτό νομίζω ότι το θέλουν πολύ στην Ευρώπη. Τώρα, ο τουρισμός ε, των ε, ποδηλατών δεν είναι μόνο δικό μου θέμα, το είπε και ο συνάδελφος Γκρός. νομίζω όμως ότι μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τα πράγματα, ειδικά για τις πολύ γειτονικέ χώρες. Ε, και εμείς στη Γερμανία κάναμε μια ένα τέτοιο μονοπάτι και πραγματικά είναι πολύ ωραία εμπειρία να πηγαίνει κανείς με το ποδήλατό του στο, στο μονοπάτι αυτό. Μάλιστα μια αποστολή ευρωβουλευτών έκανε αυτή τη βόλτα με τα ποδήλατα στο συγκεκριμένο μονοπάτι και πραγματικά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Χαίρομαι λοιπόν που και ο τουρισμός των ποδηλατών έχει μπει στο σκεπτικό μας πια, γιατί πραγματικά υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη από όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Κλείνοντα λοιπόν να πω ότι και ο τουρισμό για του ποδηλάτε ε, καθημερινά δίνει πολύ περισσότερα ε, χρήματα στου προπολογισμού από έναν ε, τουρίστα που πάει με το αυτοκίνητό του από τη μία περιοχή στην άλλη. Γιατί ο ποδηλάτη θα πάει να ψωνίσει, θα πάει στα εστιατόρια, δεν θα φύγει μέσω μια πόλη για να πάει στην άλλη. Οπότε θα βοηθήσει και την τοπική οικονομία. Να ευχαριστήσω λοιπόν και για τα εργαστήρια που οργανώσατε και στι Βρυξέλλε και στον Τάντσιχ και ο Υπουργό Νόβακ που ήταν πριν από εσά εδώ έκανε κάποιε συζητήσει με του με τους ε, συντονιστέ και είπε ότι ε, ναι, όντω έπεσε στα μέσα τη οικονομική κρίση η Πολωνική Προεδρία και είπε ότι στην Πολωνία τώρα η ε, περιφέρειες ε, θα λάβουν ε, περισσότερα χρήματα. Ε, θα ήθελα να γίνει αυτό και για τις υπόλοιπες χώρες. Εύχομαι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά. Ελπίζω και στο μέλλον και κυρίως όταν θα ξαναπάω εγώ στο Danzig να κάνω το, τη βόλτα μου με το ποδήλατο, να υπάρχουν, να υπάρχουν τα νέα μονοπάτια και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω που με βοηθήσατε όταν ήμουν παρόν στην, στην Πολωνία. Γιατί μου κάνατε τη διερμηνέα όταν το χρειάστηκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μίκαλ. Ελπίζω να υπάρξει και ποδηλατόδρομος υπερσιβηρικός. Ή μάλλον εσύ το θέλεις, Μάικλ. Κυρία Φώστρα από το ECR. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτή την πλήρη παρουσίαση που μας κάνατε. Φαντάζομαι τους τελευταίους μήνες ήσασταν πολύ απασχολημένοι. Είναι δύσκολο θέμα αυτό του τουρισμού. Και φυσικά είναι πολύ πιο ορατό τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, παρόλα αυτά παραμένει δύσκολο. Ορισμένοι έχουμε, από εμά έχουμε ανησυχίε. Ε, όταν μιλάτε για την, ε, τη νέα γραμμή προπολογισμού και για διάφορα άλλα που είπατε, ανησυχούμε. Θα σα το πω απλά. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την ορατότητα του προϋπολογισμού και γι' αυτό χρειαζόμαστε γραμμές του προϋπολογισμού, τότε αυτά τα λεφτά ε, θα πρέπει να τα πάρουμε από τομεί όπου τα λεφτά υποχρησιμοποιούνται. Δεν θέλουμε νέα γραμμή. Είναι σημαντικό τομέα, συμφωνούμε. Ε, υπάρχει μια διασύνδεση με τις μεταφορές κτλ. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρξουν επικαλύψεις δεν θέλουμε η Κομισιόν να κάνει κάτι που τα κράτη-μέλη ή οι περιφέρειες ή οι φορείς τουρισμού κάνουν. Ε, υπάρχει και ένα θέμα ανταγωνισμού επίσης. Ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε οτιδήποτε ε, και ποιος θα το προωθήσει. Έχουμε 27 κράτη-μέλη. Ποιος θα προωθήσει τι είναι το ερώτημα. Δεν θέλω να είμαι κοινική, αλλά αν δούμε το πόσες θέσεις ε, εργασίας δημιουργεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, επίσης, ε, τα πρότυπα ασφαλείας, στα ξενοδοχεία. Αν κάποιος πει, ας πούμε, ότι όλα τα ξενοδοχεία μας είναι το ίδιο ασφαλή στην Ευρώπη, αυτό είναι τεράστιο θέμα, πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που είπατε, Πρόεδρε, ε, οι σιδηρόδρομοι, τα μονοπάτια, όλα αυτά είναι σημαντικά. Επίσης, ε, αυτά που είπατε, Μάικλ, για, τα, για τους ποδηλατοδρόμους, ε, πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία είναι τα μονοπάτια αυτά, αυτοί στις λωρίδες όταν έχει ήλιο, αλλά όταν βρέχει, για φανταστείτε, κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην βρεχόμαστε. Τέλος πάντων, αυτά και καλή δουλειά. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό εδώ στην Επιτροπή μας να συζητήσουμε για τη στρατηγική του τουρισμού και είναι πολύ ευχάριστο που η κυρία υπουργό ε, είναι εδώ από μια χώρα που έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία για τον τουρισμό, για τις μεταφορές και μας, ε, έκανε την, ε, μας παρουσίασε την αναφορά της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά είμαστε μια τεράστια εσωτερική αγορά που πρέπει να έχει και κάποιες υπηρεσίες. Κυρίως όταν οι πολίτες μας θέλουν να βγούνε και λίγο προ τα έξω. Ε, πρέπει να κάνουμε τον τουρισμό μας ελκυστικό έτσι ώστε τα χρήματα να μένουν εδώ. Έχουμε πολύ ωραίε ακτέ, έχουμε εξαιρετικέ ε, υποδομές για χειμερινά σπόρα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική να τα υποστηρίζει όλα αυτά. Ενδιαφέρον επίσης ε, είναι αυτό που λέτε και για την ε, Βόρεια Θάλασσα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το πώς, ας πούμε, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την Βόρεια Θάλασσα ως έναν τουριστικό προορισμό. Ε, έχουμε τη, ε, ε, αθλητι, τουρισμό για, το, για αθλητισμό, για τα υγρά σπορ. Θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα προωθήσουμε για την εσωτερική αγορά, για να την ενισχύσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίση, κάτι άλλο να πω κυρία Υπουργέ. Στις 6 Ιουνίου ξεκινάει το Euro στην Πολωνία και στην Ουκρανία. Κάθε τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη γίνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικός σταθμός τουριστικός. Και βεβαίω η προσφορά θα πρέπει να γίνει όχι μόνο για του οπαδού του ποδοσφαίρου, αλλά όλου όσου θέλουν να επισκεφθούν την ε, ε, Ουκρανία και την ε, Πολωνία εκείνε τι ημέρε. Να συνδυάσουν λοιπόν και, την, και τον τουρισμό αλλά και την αθλητική διοργάνωση. Τι έχετε σκεφτεί εσεί για αυτό το θέμα, βεβαίω. Εμεί χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τη εθνική μα ομάδα στο Euro, προφανώ. Ελπίζω να μπορέσουμε και με τον Κλώσσα και τον Ποντόσκι να νικήσουμε. Έχουμε καταφέρει πολλά μέχρι τώρα. Ο Ποντόσκι βεβαίω στην Ντόρτμουντ ε, όταν έπαιζε με το Αμβούργο ε, έβαλε και δύο γκολ. Οπότε αυτό μας ενώνει πολύ, καταλαβαίνετε εσάς και εμάς. Το ποδόσφαιρο λοιπόν μας ενώνει και βεβαίως παίζει και έναν πολύ μεγάλο και ενδιαφέροντα ρόλο στον όλο τομέα της, ε, του τουρισμού για την ε, ανταλλαγή και την συμφιλίωση των λαών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Δεν, το, να το πει ο Πρόεδρος. Ε, ειδικά για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιρλανδία και η Πολωνία. Έχουμε πάρα πολλέ δυνατότητε να συνδέσουμε χώρε που δεν φαίνεται να, αρχικά να έχουν ε, κάποια σχέση, όπω α πούμε η Ιρλανδία με την Πολωνία. εγώ θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πολλές φορές στην πολιτική ε, κάνουμε καταγερματισμένες ε, πράξεις ή προωθούμε τον τουρισμό ή προωθούμε τις μεταφορές. Εντάξει, καλές είναι οι μεταφορές, αλλά ο τουρισμός και οι μεταφορές έχουν πολλά κοινά σημεία. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε πιο γενικά, σε πιο ευρύ επίπεδο και νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς να το προωθήσετε αυτό. Η Πολωνία έχει πολλές, έχετε μεγάλη ακτογραμμή, η Γερμανία επίσης ενδιαφέρεται για τη Βόρεια Θάλασσα ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με τις ε, προστατευόμενες ζώνες και πώς μπορούν οι, οι ε, τουρίστες να έχουν πρόσβαση και προς την Βόρεια Θάλασσα. Είναι λοιπόν ένας, είναι σημεία αυτά, μέρη, περιφέρειες που πρέπει να προστατευτούν. Οι τουρίστες ευχαρίστως πάνε στην ακτή και θέλουν να κάνουν εκεί ε, διακοπές, οπότε πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλε υποδομές μεταφορικές για να μπορούν να τους μεταφέρουν ω εκεί. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό ε, και για την στρατηγική για τη συγκεκριμένη ε, Βόρεια Θάλασσα αλλά και για άλλες, άλλα σημεία. Βεβαίω πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, αλλά πρέπει να προωθήσουμε και τον τουρισμό. Ελπίζω λοιπόν και εσείς να έχετε θέσει αυτό ως ε, βασικό σημείο έτσι ώστε να μπορέσουμε από κοινού να εκπονήσουμε μια στρατηγική. Ευχαριστώ. Και εγώ να πω, να ένα-δύο σημεία, κυρία Υπουργέ. Ένα από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης του τουρισμού είναι ο αθλητικός τουρισμός. Όπως είπε ο κύριος Κούν, ε, το ποδόσφαιρο. Αλλά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, το ράγμπι, οι υποδρομίες, ε, στην περιοχή μου, στο Λίβερπουλ, έχουμε τους μεγάλους εθνικούς ε, αγώνες υποδρομίας και έρχεται πάρα πολλοί ε, κόσμος εκεί. Ε, επίσης, Μάικλ, θα ξέρεις ότι στην βορειοδυτική Αγγλία ε, έχουμε πολλούς αθλητές που ασχολούνται με το ποδήλατο και ο αθλητικός τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και μην ξεχνάτε ότι στη Βρετανία, στην περιοχή μου μάλιστα, ε, γεννήθηκε, ε, έγινε η βιομηχανική επανάσταση. Πρέπει να υποφεληθούμε από αυτή την πλούσια κληρονομιά που έχουμε στον τομέα της βιομηχανίας, δηλαδή στα ορυχεία, τα ανθρακορυχεία, τη χαλιβουργία, τους μήλους τους εκοκιστικούς, βάμβακος. Δεν πρέπει δεν και καλά η Ευρώπη να μας υποδείξει τι πρέπει να κάνουμε. Ε, η Ευρώπη θα πρέπει να διευκολύνει τις προσπάθειες που κάνουν διάφοροι φορείς. Ε, Παραδείγματο χάρη ε, η οργάνωση μουσείων σιδηροδρόμων ή οργανώσεις των ανθρακορίχων. Θα πρέπει η οργανωσει των ανθρακοριχων θα πρεπει η ευρωπη να διευκολύνει τι προσπαθίε του, αυτού, του πόρου θέλουμε από την Ευρώπη, δηλαδή διευκόλυνση. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια ότι ζητάμε δηλαδή, από την Ευρώπη για να πάνε στον τουρισμό. Θα πρέπει η Ευρώπη να διευκολύνει τι προσπάθειε που γίνονται, ούτω ώστε να απτύξουμε έναν βιώσιμο τουρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Μια συνεργασία μεταξύ των φορέων που υπάρχουν, ε, τα ποδήλατα πούμε του του Μάικλ ή τα, οι ατμομηχανές, τα τρένα που λειτουργούν με ατμό, ε, που μου αρέσουν εμένα. Δεν θέλουμε δε και καλά τεράστια κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Εγώ όμως ε, Ξέρω πάρα πολύ καλά, ε, βρίσκομαι και σε μια άλλη επιτροπή, την Γεωργική Επιτροπή, που εκεί υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κονδύλια. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν περνάει το δικό μου κάθε φορά. Δεν, περνάνε, δεν χρηματοδοτούν τα θέματα που θέλω. Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια ε, και τους επένους προς την Πολωνική Προεδρία και να ξαναευχαριστήσω και την Επιτροπή για την πολύ επικοδομητική συνεργασία και την υποστήριξη. Αυτή είναι αναγνώριση της σημασίας που έχει ο τουρισμός στην οικονομία. Από πολλά σχόλια δόθηκε ουσιαστικά η απάντηση ότι ο τουρισμός είναι ένας οικονομικός κλάδος που εξακολουθεί να χρήση υποστήριξης προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία του και την οικονομική και την κοινωνική. Γιατί είναι σημαντική ε, η η συμμετοχή του τουρισμού στο κοινωνικό ΕΠ Αυτή τη στιγμή είναι 5% στο κοινωνικό ΕΠ, συνεχώς όμως αυξάνεται και θα πρέπει να διαδώσουμε αυτή τη ε, γνώση για τη σημασία του τουρισμού. Και όλες ε, οι βάσεις που σας είπαμε ε, στηρίζονται και στα στοιχεία από δορυφόρο, που είναι πολύ σημαντικά Καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε μια κοινή ενιαία βάση στατιστικών δεδομένων για το τουριστικό δυναμικό. Η ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης είναι απείρως ε, σημαντική και χρήσιμη και για να στηρίξουμε τον ε, τουρισμό, αλλά και για να βοηθήσουμε όλους τους επίδοξους επιχειρηματίες να διεκπαιρώσουν τα σχέδιά τους και σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Πολλές ε, παρατηρήσεις μίλησαν ε, για τον αηφόρο τουρισμό. Κατά τη γνώμη μου, ο αηφόρος τουρισμός είναι από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της νέας ανακοίνωσης. Και όλες οι νέες πρωτοβουλίες που αναφέρονται, για τα, που αναφέρονται στα ευρωπαϊκά μονοπάτια, είτε είναι πεζοπορικά, είτε ποδηλατικά, είτε είναι μονοπάτια πολιτιστικής κληρονομιάς ή βιομηχανικής κληρονομιάς, όλα αυτά οι πρωτοβουλίε για τέτοιου είδου μονοπάτια χρήζουν υποστήριξη. Κάποιο ρώτησε πώς θα προαγάγουμε την Ευρώπη, πώ θα στηρίξουμε αυτή την προβολή και την προαγωγή τη Ευρώπη και των πολλών σημαντικών αξιοθεάτων τουριστικών που διαθέτουμε. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά μονοπάτια, τα ευρωπαϊκά ίχνη και νομίζω ότι αυτό είναι που μας ενώνει. Γι' αυτό και το σχέδιο της προώθησης ε, του, της Ευρώπης ως, ευρωπαϊκού, του προορισμού, ως τουριστικού προορισμού στις τρίτες χώρες, η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή του Τουρισμού έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να, να διαφημιστούμε από κοινού ε, τα, τα κράτη-μέλη που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα της Ευρώπης ως συνόλου. Να δημιουργήσουμε κάποιες κοινέ τουριστικές προσφορές, και κοινά τουριστικά προϊόντα και μονοπάτια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Βαλτική θάλασσα ή τη νέα πρωτοβουλία ε, για τις 50.000, ε, τους 50.000 τουρίστες που είπαμε. Εδώ θέλουμε να εκπονήσουμε κάποια κοινά προϊόντα, όχι μεμονωμένα κρατικά τουριστικά προϊόντα και τουριστικές προσφορές. Αυτό που αναζητούμε είναι κάποιοι εταίροι για να δημιουργήσουμε κοινά προϊόντα, πολωνολιθουανικά, πολωνογερμανικά, στα πλαίσια της ομάδας του Βίσεγκρατ προϊόντα τουριστικά του Βίσεγκρατ. Κατά τη γνώμη μου τέτοιου είδους κοινά προγράμματα και σχέδια ε, έχουν ε, πολλές πιθανότητες να ευοδοθούν, γιατί θα είναι και πιο ανταγωνιστικά και μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή των εξοκοινωτικών τουριστών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μου διέφυγε στην προηγούμενη μου παρουσίαση, που παρέλειψα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών παρουσιάστηκε μια πρωτοβουλία και λήφθη η απόφαση ώστε εκπρόσωπο τη ε, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι μόνιμο προσκεκλημένο στα άτυπα Συμβουλία Υπουργών Τουρισμού. Αυτό σε μεγάλο βαθμό διευκολύνει την ροή των πληροφοριών μεταξύ Συμβουλίου και της Επιτροπής σας. Και έτσι μπορούμε από κοινού να λαμβάνουμε πραγματικά σημαντικές αποφάσεις για τα θέματα του ευρωπαϊκού τουρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση. Βέβαια, οι διαπραγματεύσει για τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ για την περίοδο 2013-2020 θα απαιτήσουν πολλού συμβιβασμού. Έχω πάντως την αίσθηση ότι λαμβάνοντας υπόψη αυτό το τεράστιο δυναμικό που έχει ο τουρισμό για την ευρωπαϊκή οικονομία, θα πρέπει να δώσουμε στον τουρισμό τη θέση που του αξίζει. Ίσως όχι μέσω ενός ξεχωριστού χρηματοδοτικού μέσου, αλλά να δώσουμε στον τουρισμό τη θέση που του αξίζει στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής. Αυτό συνδέεται και με μία ερώτηση ε, για τα όρια, τα εμπόδια, τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε ε, ε, σε ό,τι αφορά την έκθεση του κυρίου Φιντάντζη. Θα ήθελα να πω ότι η υλοποίηση όλων αυτών των νέων πρωτοβουλειών για, τη, για τον τουρισμό και μάλιστα μετά τη θέση και της συνθήκης Λισαβόνας συνέπεσαν με μια πολύ αρνητική συγκυρία με πολύ ε, αντίξωες συνθήκες και οικονομικές ε, και χρηματοπιστωτικές. Στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας είχαμε την ηφαιστιακή τέφρα, την έκρηξη του ηφαιστείου και άρα την, τον εγκλωβισμό και την, ε, τον εγκλωβισμό ε, χιλιάδων Ευρωπαίων τουριστών στα αεροδρόμια που έμειναν καθυλωμένοι γιατί δεν μπόρεσαν να βάλουν τις πτήσεις τους. Όλες αυτές, ε, όλα αυτά τα γεγονότα ήταν πολύ σημαντικά και δυσκόλεψαν ε, και την Προεδρία. Πάντως όλες οι προτεραιότητες και για τον αηφόρο τουρισμό είναι σημαντικό να προωθηθούν και να υλοποιηθούν. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να προωθήσουμε τον τουρισμό και να τον διαφυλάξουμε και στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα των επιβατών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, για την οδηγία 313 ε, που είναι πολύ σημαντική από άποψη τουρισμού. Το 2010 είχαμε την ε, την κρίση και σίγουρα η κρίση αυτή θα τροποποιήσει το, την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Θέλουμε οπωσδήποτε πάντως να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών και των καταναλωτών. Ο τουρισμός είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση και με τις μεταφορές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το χαρτοφυλάκιο σας καλύπτει και τον τουρισμό. Όταν μιλούμε για ε, τουρισμό δεν μπορούμε να ξεχνούμε τις μεταφορές, γιατί με τις συγκοινωνίες μετακινούνται οι τουρίστες. Και μάλιστα για την Πολωνία έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα αυτό. Θέλουμε με τη βελτίωση των οδικών μας ε, υποδομών των οδικών, να καταστήσουμε πιο ελκυστικές τις πολωνικές περιφέρειες και πιο προσιτές για τους τουρίστες. Και σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την ε, Βαλτική θάλασσα, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε συνεχώς επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών, που εξασφαλίζει το συντονισμό των εργασιών για το έγγραφο αυτό και τη στρατηγική αυτή και θα τη στηρίξουμε ε, και στα πλαίσια των άλλων τουριστικών πρωτοβουλειών, τη στρατηγική για τη, για τη Βαλτική. Σε ό,τι αφορά τώρα την βιομηχανική κληρονομιά και για την Πολωνία, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο ε, τουριστικό προϊόν, γιατί η νότια περιοχή της ε, χώρας μας στηρίζεται στην αξιοποίηση τέτοιων υποδομών, ε, ιδιαίτερα των ορυχείων, και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα εγκαταλειμμένα ορυχεία για τουριστικούς σκοπούς. Μάλιστα είχαμε ένα διαγωνισμό ε, εντέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να αξιοποιηθούν ε, μεταβιομηχανικά αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και μάλιστα στο Κατοβίτσε είχαμε τη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Επιτροπής Τουρισμού που ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με τον βιομηχανικό τουρισμό. Γιατί και χάρη στο βιομηχανικό τουρισμό μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε κάποια ευρωπαϊκά μονοπάτια της βιομηχανικής μας κληρονομιάς και να τα προωθήσουμε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τον αθλητισμό. Ε, ο, ο τουρισμός ε, στην Πολωνία εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού. Οπότε συνδυάζονται τα δύο θέματα. Φυσικά είμαι υπέρ ε, των διατάξεων της νέας ανακοίνωσης για την πρόθεση αθλητικών ε, εκδηλώσεων ε, και την ανάδειξη του τουρισμού και του αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα το επικείμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πολωνία, σίγουρα έχουμε χάρη στο πρωτάθλημα αυτό μεγάλη ευκαιρία διαφήμιση και προβολή τη χώρα μα, όχι μόνο από τουριστική άποψη, αλλά και από οικονομική και από πολιτιστική άποψη. Ευελπιστώ ότι θα πετύχουμε σε αυτέ τι εξετάσει. Και ελπίζουμε ότι όσοι θα μας επισκεφθούν στο διάστημα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου θα ξαναγυρίσουν στην Πολωνία και μετά από αυτό. Και μάλιστα ε, με λίγου μήνε μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πολωνία, θα έχουμε του Ολυμπιακού στο Λονδίνο, που είναι νομίζω η σημαντικότερη παγκοσμίω αθλητική εκδήλωση οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Είναι εξαιρετικό αθλητικό γεγονό. Αλλά για όλε τι χώρε ε, που συμμετέχουν σε τέτοιου είδου αθλητικέ εκδηλώσει, ε, η συμμετοχή του και μόνο είναι ένα είδο προβολή. Βέβαια, Έχουμε στα επόμενα χρόνια και άλλες τέτοιες ε, εκδηλώσεις. Ε, θα φιλοξενήσουμε ε, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ και φυσικά και το Πρωτάθλημα Handball. Ελπίζω να έχουμε σημαντικές επιτυχίες. Και αυτά κύριε Πρόεδρε, από πλευράς μου να σας ξαναευχαριστήσω θερμότατα για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε και ευελπιστώ ότι και στο μέλλον ο τουρισμός μπορεί να υπολογίζει στη δική σας υποστήριξη. Εμείς ε, σίγουρα θα συνεχίσουμε την προσήλωσή μας στην υλοποίηση όλων αυτών των σχεδίων και πρωτοβουλειών και εύχομαι καλή τύχη και στη Δανική Προεδρία και στην επόμενη την Κυπριακή και ελπίζω να συνεχίσουν με δραστήριο τρόπο την ε, προώθηση και υλοποίηση όλων αυτών των πρωτοβουλειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σοβιεράισκα. Σας ευχαριστούμε και για την επισκόπηση που μας κάνατε. Και για τις απαντήσεις που δώσατε στους ευρωβουλευτές. Καλή τύχη στο μέλλον για στα πλαίσια των εργασιών σας ως Υπουργός Τουρισμού της Πολωνίας.